Καλημέρα, θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια δεύτερη. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν ε, επιθυμίες αλλαγής. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι εγκεκριμένη. Γνωρίζετε ποιε είναι οι γλώσσες στην οποία υπάρχει διερμηνία, υπάρχει web stream για όλη την συνεδρίαση. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Ο κύριος Μαρτσάτ. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με την ημερήσια διάταξη. Αύριο υπάρχει η ακρόαση για την υπόθεση Σαλμάιερ. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είχε προβλεφθεί 2,5 με 4,5 και 4,5 με 5,5 θα υπήρχε η ανταλλαγή απόψεων για το ψήφισμα. Αυτό το δεύτερο σημείο, δηλαδή 4,5 με 5,5 θα μπορούσε να συντομευθεί λίγο, γιατί μόλις θα έχουμε δει το κείμενο. Έχω την εντύπωση ότι ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε λίγο και για αυτά που μας είπε ο κύριος Έτιγκερ για να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για την ακρόαση. Δηλαδή 10 λεπτά για το θέμα αυτό φτάνει έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για τον κύριο Ατίνγκερ. Προς το παρόν δεν ξέρουμε αν θα έχει περισσότερο χρόνο από τη μια μισή ώρα που αρχικά μας έχει διαθέσει. Α, νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό το χώρο. Ελπίζω να υπάρξουν πολλές ερωτήσεις, να μπορέσει να απαντήσει σε αυτές και ελπίζω ότι μέχρι αύριο θα υποβληθεί ένα σχέδιο κειμένου. Να δούμε και οι συντονιστές. Ε, εγώ πολύ θα χαρώ να υπάρξει η υποστήριξη. Το κείμενο αυτό, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ποια είναι τα μαθήματα που μπορούμε να αποκομίσουμε και βεβαίω πώ μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τώρα, το σχέδιο κειμένου το αργότερο αύριο το πρωί θα είναι έτοιμο και θα το έχετε. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι φυσικά μπορείτε να υποβάλλετε και τροπολογίες. Είτε δηλαδή το υπογράψετε είτε όχι το κείμενο. Μαρτίνα. I think that it sounds very reasonable Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λογικό είναι αυτό που προτείνει ο Μπαρτ Στάιφ. Γιατί για μας είναι σημαντικό να έχουμε χρόνο για να θέσουμε τις σωστές αρετήσεις. Αν δείτε λοιπόν ότι ο καλεσμένος μας έχει πιο πολύ χρόνο τότε, να το σκεφτούμε για να έχουμε περισσότερο χρόνο ακρόασης και χρόνο για ερωτήσεις και να τα συμπυκνώσουμε περισσότερο αυτά τα του ψηφίσματος. Εάν μπορείτε λοιπόν, θα ήταν πολύ καλό. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν στον Εμποδίο Επίτροπο, αν μπορεί να μας αφιερώσει περισσότερο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να συζητήσουμε για το σχέδιο κειμένου, το σχέδιο ψηφίσματος. Ε, θα βρεθεί χρόνος να γίνει μέχρι τις ε, 4,5. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν δούμε ότι χρειαζόμαστε λιγότερο χρόνο για το άλλο ψήφισμα, που είναι απλώς μια γνωμοδότηση. Κοιτάξτε, αύριο το πρωί έχουμε και το θέμα της Ογκαρίας και κάποια άλλα θέματα. Ο κύριος Φάνιγεν. Ε, ναι, θα συμφωνήσω όμως με τους προηγούμενους ομιλητές. Ε, den Haushaltskommissar an. Und dann ist klar, dass wir natürlich viele Fragen. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς ε, ελπίζω να υπάρξουν πολλές ερωτήσεις. Θα κάνω εγώ μια πρώτη παρουσίαση. Η, εδώ, η ομιλία του, μετά οι συντονιστές, ε, κατόπιν ε, μια σειρά ομιλητών. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουν να θέσουν τις ερωτήσεις τους και οι συντονιστές, αλλά βεβαίως και όλα τα μέλη ελπίζω να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Δύο-τρία λεπτά χρόνος ομιλίας για τον καθένα νομίζω ότι αρκεί. Το λόγο έχει ο Μπάρτα. Αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί με το χρόνο και μιλήσουν και οι συντονιστέ, θα πρέπει να γίνει ερώτηση-απάντηση προ τον κύριο Έτιγκερ, σαν πινκ-πονγκ. Αυτό έχετε προβλέψει ή να απαντήσει καλή, μια και καλή ο κύριο Έτιγκερ όλες τις απαντήσεις. Νομίζω ότι αν το κάνουμε ένα-ένα, ερώτηση και απάντηση, θα είναι πιο ζωντανή η συζήτηση, πιο ενδιαφέρουσα. Διότι ξέρουμε ότι πολλές ερωτήσεις δεν θα απαντηθούν στο τέλος αν τις απαντήσω όλες μαζί ή μπορεί να έχει και την ευκαιρία να αποφύγει κάποιο. Γι' αυτό λοιπόν θα προτιμούσα την ε, μορφή του ping πόνγκ. Έτσι έχουμε προβλέψει ακριβώς στο το παρόν τουλάχιστον. Ναι, να κάνουμε αυτό του είδους ε, ερωτήσεις-απαντήσεις Δύο λεπτά, τρία λεπτά απάντηση του Επιτρόπου. Έτσι το έχουμε σκεφτεί έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποια χρονικά πέντε λεπτά, ας πούμε, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος. Και τώρα περνάμε στο τρίτο σημείο της ημερησίας διάταξης, συζήτηση ο κύριος Σέλερ. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε συζητήσει τόσο πια για αυτό το θέμα, το έχουμε κάνει και ακροάσεις, ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε και να φτάσουμε στην τελική φάση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Απλώς να σας ενημερώσω ότι θα αποσύρω την τροπολογία 421. Έχουμε βέβαια συζητήσει με τη γραμματεία γι' αυτό, το έχουμε προσπαθήσει να βρούμε λύση. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, αλλά τώρα ε, αποσύρουμε την τροπολογία 41. Genau, 36. Σελίδα 36 της ψηφοφορίας. Ωραία, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ελέγχουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Πιέστε το κουμπάκι σας για να δούμε αν λειτουργούν όλα. Υπάρχει κάποιος που έχει ξεχάσει την ε, κάρτα του. Όχι. Κάποιος λείπει. Εντάξει, όλοι ψήφισαν. Δεν υπάρχει κανείς που περισσεύει για την απαλλαγή 1, 2, 3. Θα ψηφίσουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 16 πέρα 7 κατά εγκρίνεται. Τελείωσε λοιπόν το θέμα αυτό, προϋπολογιόλος μας επιτροπής. Και τώρα πετάμε στην απαλλαγή... Α, όχι, των ε, διαφορετικών τελευταίων υπηρεσιών. Αυτό έχει γίνει. Κλείσιμο των λογαριασμών. Αυτό πρέπει να το ψηφίσουμε. 11, 22 τροπολογία υπέρ. 22 υπέρ κατά αποχέας. Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 22. Τέλος. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Προφορική. Υπάρχει κάποιος που είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Υπάρχουν. Άρα απορρίπτεται η προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσει. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο με ξεχωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα υπέρ. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το 32 παρακαλώ ελέγχουμε. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. 33 σε 5 τμήματα. Ένα. Υπέρ εγκρίνεται. Δύο το δεύτερο τμήμα. Αποχές απορρίπτεται και αυτό. Τρίτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε το τέταρτο τμήμα. Νομίζω απορρίπτεται. Ναι, ναι, ναι, απορρίπτεται. Πέντε, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 με προφορική. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Απορρίπτεται η προφορική. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. δύο, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ευχαριστώ πολύ. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Α, συγγνώμη, το 37. Ελέγχουμε. 37. Δύο συνάδελφοι δεν ψήφισαν. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 με προφορική δεν υπάρχουν αντιρρήσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 με προφορική χωρίς αντιρρήση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 50 με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 με προφορική τροπολογία χωρίς αντιρρήσεις υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 52. ...52 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. 53. Κατά αποχές. Α, ελέγχουμε την 53. Τέλος απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά ελέγχουμε την 58.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 67 κατά πέπτη, 69 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 69, νομίζω ότι απορρίπτεται. 69. Τέλος, εγκρίνεται, Κάνω, έκανε λάθος. 70 υπέρ κατά αποχές. 70 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 71. 71. Τέλος. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 74 και 75. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. 78 νομίζω ότι η διαφορά είναι μία ψήφος. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά Αποχές υπέρ, 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 με προφορική τροπολογία. Έχετε αντίρρηση. Ε, ωραία. Μόνο την 81 λοιπόν, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Είναι ταυτόχρονα με την 80, με προφορική τροπολογία η 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 με προφορική υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 82. Τέλος, εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά, αποχές, 83 και 84 ελέγχουμε ηλεκτρονικά και τις δύο μαζί. Τέλος. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Όχι, να ελέγξουμε την 86. Τέλος. Απορρίπτεται. Είναι σημαντικό να ελέγχουμε. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ. Κατά. Όχι, κατά πίπτη 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε την 95. Τέλος, εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 98. Κατά πίψη. 99 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 ελέγχουμε. Τέλος, εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 109. Και περνάμε στην 110 υπέρ εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ με προφορική, χωρίς αντιρρήσεις, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 118 ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται ξεκάθαρα. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120. Που ταυτίζεται με την 121-122 αποσύρθηκε υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 125 με προφορική χωρίς αντιρρήσει υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 124 υπέρ Α, πάμε στην 24-23 κατά πίπνο, 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά Ελέγχουμε. 127. Έχω την αίσθηση ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να βεβαιωθούμε. Αυτή η χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει στο να σηκώνετε τα χέρια ε, ε, δημιουργεί προβλήματα. Εγκρίνεται, ναι. 128 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 135 δεν θα υπάρξει ψηφοφορία. 136 ε, υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά εποχές 139 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος, απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται απορρίπτεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 146 και 147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 148 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 150. Τέλος, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 161. 161 ελέγχουμε. Πέρας εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 164. Τέλος. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166 δεν υπάρχει ψηφοφορία. 167 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά απο... αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 αποσύρθηκε 179 με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά να ελέγξουμε. 180 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε και αυτό. Ψηφίζουμε για την 181. Απορρίφθηκε. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 αποσύρθηκε. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188. Καταπίπτει 190 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε για να σιγουρευτούμε. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 193. Απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197 αποσύρθηκε, 198 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 201 δεν ψηφίζουμε, 202 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά έχουμε προφορική τροπολογία, χωρίς αντιρρήσεις, για το ίδιο το κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε. Έχω την αίσθηση ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να βεβαιωθούμε. Ναι. Υπάρχει αυτή η χρονοκαθυστέρηση κάθε φάση της προφορίας. Ναι, εγκρίνεται πράγματι. 205 υπέρ, κατά, αποχές.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 εγκρίνεται. 218 αποσύρθηκε. 219 με προφορική τροπολογία χωρίς αντιρρήσεις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 220 με προφορική τροπολογία χωρίς αντιρρήσεις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά αποχές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 Ψηφίζουμε επί της 226. Ε, One green too much. One green too much. Ένας υπεράριθμος από τους πράσινους. Yeah. Okay, thanks. Yeah, okay. Yeah, genau. Das ist abgelehnt. Ακριβώς, ωραία. Απορρίφθηκε. 227 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 228 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 229 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 230 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 230 ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Yeah, check is over. Clearly rejected. Τέλος. Απορρίφθηκε. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 233 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 232. Ψηφίστε παρακαλώ. Ναι. Απορρίφθηκε. 200... 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 237 παρακαλώ. Yeah, Ναι, απορριφθήκε. 238 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 240 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.41, 42, 43 υπέρ, κατά αποχές, να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. 241 έως 43 εγκρίνονται. 2.44 και 45 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε και αυτό καλύτερα. Ψηφίζουμε επί των τροπολογιών 2.44-2.45 ηλεκτρονικά. Das Εγκρίνονται. 246. Καταπίπτει. 247 καταπίπτει. 248-249 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. This you can believe me because 48 49 Check. Ψηφίζουμε επί των τροπολογιών 248-249 ηλεκτρονικά. It is rejected. Απορρίπτονται. 2.50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.51, 2.52 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτονται. 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.54 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 2.55 και 56 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε καλύτερα. Για να είμαστε σίγουροι, ψηφίζουμε στροπολογίες 2.55-2.56 ηλεκτρονικά. Εγκρίνονται. 2,57 υπέρ. Καταπίπτει 2,57. Προφορική τροπολογία χωρίς αντιρρήσεις υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2,58, 2,59, 2,60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε καλύτερα σας παρακαλώ. Ηλεκτρονικά ψηφίστε. Τέλος της προφορίας εγκρίνονται. 2.61 έως 2.66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 2.67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.68 έως 2.71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ας το ελέγξουμε. 268 έως 271. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος, εγκρίνεται. Συγγνώμη και σας ευχαριστώ που ζητήσατε τον έλεγχο. 273-74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Θέλετε να ελέγξουμε. 272-273 ψηφίζουμε τώρα. Τέλος. Εγκρίνονται με μία ψήφο διαφορά. Ευχαριστώ. 2.74 αποσύρθηκε, 75-76 υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα και αυτό. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για τις 275 2.75-2.76. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Εγκρίνονται. Με μία ψήφο διαφορά. 277-278 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε και αυτό. Σας παρακαλώ ψηφίστε επί των τροπολογιών 277-278. Τέλος, εγκρίνονται. 279 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 279. Τέλος, απορρίπτεται. 281 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη. 281. 281. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. No, no, no. 79 was adopted. Η 279 εγκρίθηκε. 279 was rejected. Απορρίφθηκε, συγγνώμη. 200... Where are we? 280, I'm sorry. 200... Έχετε δίκιο, συγγνώμη. 280 υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε, σας παρακαλώ. 280. Ψηφίζουμε για τροπολογία 280. Απορρίπτεται. 281. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 281. Αν θέλετε να το ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα της 281. Εγκρίνεται. 282 με προφορική. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 283. 282. Ναι, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 282. Ψηφίστε παρακαλώ. Yeah. Yeah. 283 to 285 in favor. 283-285 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 286 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 2.87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.91 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε σας παρακαλώ να είμαστε σίγουροι. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 291. It is adopted. 29. Εγκρίνεται. 293 υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να το ελέγξουμε σας παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ για την ε, τροπολογία 293. Τέλος, απορρίπτεται. 294 υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε σας παρακαλώ ψηφίστε για την 294. It is rejected. Απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά σας παρακαλώ συνάδελφοι. Ψηφίστε επί της τροπολογίας 296. Εγκρίνεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 300 δεν ψηφίζουμε, 301 υπέρ κατά αποχές Μπορούμε να το ελέγξουμε σας παρακαλώ. Ψηφίστε για την τροπολογία 301. It is Εγκρίνεται. 302 υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε σας παρακαλώ συνάδελφοι. Ψηφίστε για την τροπολογία 302. Εγκρίνεται. 303 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 304 αποσύρθηκε, 305 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 306 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 307 αποσύρθηκε, 308 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, ας το ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Όχι, εγκρίνεται, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Ναι, ναι, εγκρίνεται. 309 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 310 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 311 υπέρ, κατά αποχές μπορούμε να το ελέγξουμε σας παρακαλώ νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να βεβαιωθούμε όχι σαφώς μάλιστα απορρίφθηκε 312 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 313 με προφορική τροπολογία συγγνώμη τι 312 ωραία ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 312 ελέγχουμε την 312 Απορρίφθηκε. 3.13 με προφορική τροπολογία χωρίς αντιρρήσεις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την 3.16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.20 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 3.21 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 3.22 υπέρ, κατά, άποχες, Μπορούμε να το ελέγξουμε. Σας παρακαλώ ψηφίστε για την τροπολογία 322. Εγκρίνεται. 3.23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.24 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να το ελέγξουμε σας παρακαλώ. Ψηφίστε για την 3.24. It is adopted. Εγκρίνεται. 3.25 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 3.26 καταπίπτει. 3.27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 328 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 329 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 330 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 331 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε σας παρακαλώ. 331. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το δούμε καλύτερα. Όχι, απορρίπτεται. 3.32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.34 υπέρ, κατά, αποχές, μπορούμε να το ελέγξουμε. 3.34, ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 3.35 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε σας παρακαλώ. Ψηφίστε για την 335. It is rejected. Απορρίπτεται. 336 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 337 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 338 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 339 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.41 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε, νομίζω ότι εγκρίνεται. 3.40 3.41 με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. 3.41, 3.41. Εγκρίνεται. 3.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.43 κατά πίπτη. 3.44 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 3.44. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Απορρίπτω. 3.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 346 με προφορική τροπολογία χωρίς αντιρρήσει. υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 3.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. 49 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 3.49 όχι σε δύο τμήματα απλώς αν απορρίπτω η προφορική τροπολογία εγκρίθηκε 350 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 351 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 352 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 353 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 354 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε για την 354. Απορρίπτεται 355 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται. 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 366 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 365 καταπίπτει. 367 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 369 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε 369 Εγκρίνεται. 3.70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.73 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. 3.73. Μα λείπει μια ψήφο, αλλά απορρίπτεται. 374 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. 377. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ναι, εγκρίνεται. 378 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 381 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 382 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 383, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 384, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε. 384. Εγκρίνεται. 385. Καταπίπτει. 386. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 387. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 388. Υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται. 389 με προφορική τροπολογία δεν υπάρχουν αντιρρήσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 390 υπέρ κατά Α, Καταπέμπτει ένα εγκριθεί προφορική. 390 και 391. Τι ψηφίζουμε. 392. Ε, Καταπίπτει επίση 3,93 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 3,94 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 3,95 και 96 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνονται. 3,97 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 3,98 υπέρ. Κατά αποχέ ε, απορρίπτεται. 3,99 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 400 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 401 δεν ψηφίζεται. 402. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 403. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 404. Υπέρ. Κατά αποχέ. Νομίζω ότι απορρίπτεται ελέγξουμε 404. Απορρίπτεται. 405. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 406. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 407 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 409 ναι. 408 έλεγχος. Απορρίπτεται, ευχαριστώ που ζητήσατε έλεγχο. 409 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 410 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 411 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 413 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 414 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, να ελέγξουμε 414. Απορρίπτεται. 415 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 416 δεν ψηφίζεται. 417 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 418 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ναι, εντάξει να ελέγξουμε το 418 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. αυτέ τι δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 419 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 320 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 421 21 αποσύρεται 422 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 424 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 425 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 426 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 427 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ, να ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα 427. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα 427 υπέρ κατά αποχές 428 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 429 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 430 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 431 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 432 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 433 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 433 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 435 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 436 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 438 με προφορική τροπολογία δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Να ελέγξουμε την προφορική. Το ίδιο το κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 439 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε για την 439. Απορρίπτεται. 440 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 441 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 442 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 443 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 434, 444 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 445 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 446 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 447 υπέρ Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά να ελέγξουμε 447. Εγκρίνεται. 448 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 449 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 450 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άθετ 1 ω 5 on block. Άθετ 1 ω 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8. Άφετ 8 ως 11 unblock. 8 ως 11 άφετ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Δέδε 1 έως 4 unblock. 1 έως 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 5. Δεβε 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύ 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύ 9. Καλύπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Μπορούμε να ελέγξουμε για την 11. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 1 ως 6 unblock. 1 ως 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 9. Έμπλ 9 έως 12 Εντάξει λοιπόν, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές καλύπτεται. Και η 11. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV1 έω 5 unblock. NV1 έω 3 unblock υπέρ. Καλύπτονται, δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε. NV4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 έλεγχος. Πέρας, απορρίπτεται. Η NV2 δεν καλύπτεται. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την απαλλαγή της Επιτροπής. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί δεν έχουν καμία σχέση με την απαλλαγή της Επιτροπής. Όχι, κανονικά δεν ψηφίζουμε διότι είναι εκτός πεδίου, εκτός θέματος. NV6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. 14, 14 και 15 καλύπτονται, 16 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε για την 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. NV17. Μερική απαλλαγή. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Τραν 1. 1. Ε, υπέρ κατά εποχές ε, εγκρίνεται 4, καλύπτεται 5 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 καλύπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά εγκρίνεται 11, καλύπτεται 12, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14, υπέρ κατά καλύπτεται ωραία και 15, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17, υπέρ 18, ε, υπέρ, 19 μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20, υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε εγκρίνεται. 21 καλύπτεται, Ρέτζι 1 έως 3 καλύπτονται, 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ, κατά να ελέγξουμε. απορρίπτεται 6 και 7 καλύπτονται 8 υπέρ κατά αποχές <laughs> γκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα καλύπτονται άγκρι. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Από, ε, 4 υπέρ. Κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε για την άγκρι 4. Άγκρι 4. Άγκρι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την άγκρη 6. Εγκρίνεται 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8, μάλλον 12 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει πλειοψηφία. Ναι, εγκρίνεται. 13 καλύπτεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για το 17. Ίσως να υπάρχει πλειοψηφία. Ναι, οι υπόλοιπε άγκροι καλύπτονται. Πες 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5, πες 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 8 Εδώ στον κατάλογο μου έχει αρνητικό πρόσημο. ΠΕΣ 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε για τη 10. Έμεινα άναυδη, γι' αυτό ρώτησα τι συμβαίνει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. 11 καλύπτεται. Κουλτ 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 4, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα θέλω να είμαι σίγουρη. Απορρίπτεται. Ξεκάθαρα. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ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 Κουλτ 12 έως 17 καλύπτονται. 17 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε για την Κουλτ 17. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ 1 υπέρ κατά να ελέγξουμε για τη φαμένα. Είναι υπεράριθμοι οι βουλευτέ του ΕΛΚ. Όχι. Ωραία. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές να ελέγξαμε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Ε, 7 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την ΦΑΜ 7. εγκρίνεται με διαφορά. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το ψήφισμα συνολικά με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται αυτή. Πέρας 18 προς 4 συγχαρητήρια στον εισηγητή. Yeah, absolut. Tolle Leistung. So. I put to the vote the discharge special reports of the Court of Auditor. Τώρα περνάμε στο θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου, απαλλαγή, δική έκθεση. Έχετε σχόλια, όχι. Τροπολογία 1, υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ κατά εγκρίνεται. 3, υπέρ κατά εγκρίνεται. 4, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 7 7 ηλεκτρονική ψηφοφορία 7. Τέλος της ψηφοφορίας. Υιοθετείται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 10. 10. Τέλος. Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 13. 13. Τέλος, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται, 15 16 υπέρ κατά 17 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 17. 17. Τέλος. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 21. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές. Ψηφίζουμε την 21. 21. Τέλος. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Ευχαριστώ πολύ. 18 υπέρ, 3 κατά. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα ψηφίζουμε την ε, έκθεση όσον αφορά τον έλεγχο των ε, οικονομικών και χρηματοπιστικών δραστηριοτήτων για την ΕΤΕΦ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και να δούμε πώς θα πάει η ψηφοφορία. Ίσως αλλάξω σχόλια μετά. Όχι, όχι. Είστε έτοιμοι. Ένα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 6. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές. Α, συγγνώμη, ξέχασα τη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 19 νομίζω εγκρίθηκε τέλος ναι εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά 21 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία 24. Απορρίπτεται 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 26. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και την 27. 27. Απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ 29 υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται αλλά να ελέγξουμε την 29 ηλεκτρονικά εγκρίνεται 30 υπέρ υπέρ της 30 κατά αποχές ελέγχουμε την τροπολογία 30. Εγκρίνεται. Η 31 αποσύρθηκε, 32 υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε την τροπολογία 32. Τέλος. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Συμβιβαστική 5 εγκρίθηκε 39, απορρίφθηκε 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε 41 υπέρ, κατά, αποχές,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 τρία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και η 65 εγκρίθηκε. 64 υπέρ κατά αποχές. Α, το πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα του 64, της τροπολογίας 64. ηλεκτρονικός έλεγχος. Το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε με σαφήνεια. Το δεύτερο απορρίπτεται σαφέστατα. 65 εγκρίθηκε, συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε, 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 69. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι η 68 καταπίπτει η 71 και η 72 επίσης. Η 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 1 υπέρ κατά αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την Ίντα 1. Εγκρίνεται. 2 με 6. 2 με 6 unblock. Ίντα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές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 Και τώρα με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Εγκρίνεται 20 υπέρ, 3 αποχές, 0 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ψηφίζουμε τώρα την ε, έκθεση του κυρίου Παντιό. Θέλει ο συγητής να πάρει το λόγο. Όχι. Ξεκινάμε με την τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 15 Τέλος, απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. αγκρίνεται.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 Προφορική 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47. Καταπίπτει. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 52. Εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 55 νομίζω ότι απορρίφθηκε. απορρίφθηκε. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 56. Έλεγχος 56. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την τροπολογία 67. Εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 71. 71. Εγκρίνεται. 72 το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το 73 δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται νομίζω. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 77. Δεν είναι εύκολο. Εγκρίνεται. Ένα υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε την ένα. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τροπολογία. Τέσσερα. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται.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 κατά Λιμπένα το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα της Λιμπένα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε χωρίς νούμερο. Το δεύτερο τμήμα του 1 καλύπτεται. Λίμπε 2 καλύπτεται. Καλύπτεται το 2 του Λίμπε. 3 υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. Λίμπε 4 υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. 5 καλύπτεται. Στη δική μου λίστα καλύπτεται. Το 5 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 6 καλύπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 8 πρώτο τμήμα καλύπτεται. Λίμπε 8 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα λοιπόν, το σύνολό του αρχής της ψηφοφορίας, τέλος 21 υπέρ Μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τέλος των ψηφοφοριών. Και θα προετοιμάσουμε τώρα την αποστολή μας στη Λετωνία και τη Λιθουανία. Yeah. Please. Παρακαλώ αποχωρήστε ήχος. So. So. Ich rufe Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης.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 Λοιπόν, πάμε. Προετοιμασία αποστολή στη Λετωνία και τη Λιθουανία. 3 έω 6 Απριλίου. Πήραμε και μια μέρα παράταση και δυστυχώ μόνο τρει από εμά θα πάμε. Και τρει καλά θα είναι. Δύο να μην είμαστε. Είναι κρίμα πραγματικά. Γιατί νομίζω δεν έχουμε ε, ε, επισκεφτεί ποτέ τη Λετωνία. Και δεδομένων και των προβλημάτων και στον τραπεζικό κλάδο είναι κρίμα. Πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε με αυτή τη χώρα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Τη Λιθουανία την έχουμε ασχοληθεί. Αυτή είναι μια follow-up ε, αποστολή. Θα πάμε στον πυρηνικό αντιδραστήνα στο Ιγναλίνα και θα ελέγξουμε και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις εργασίες εκεί και η προηγούμενη αποστολή μας αυτό έχει ως θέμα και τώρα το θα εξετάσουμε βεβαίως και αιτήματα ε, για νέα χρηματοδότηση υπό το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω στους συναδέλφους από την Επιτροπή Αποσχόλησης. Θέλουμε να ακούσουμε τι θα, τι θα κάνουμε εκεί. Θα ξεκινήσουμε ε, Έχουμε και εκπροσώπους της Γενικής ε, Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής. Κύριε Κολέζα, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, DG Radio. Θα επισκεφτείτε λοιπόν μια σειρά από έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαφορετικά Επενδυτικά Ταμεία στη Λετωνία και κάποια αντίστοιχα έργα στη Λιθουανία. Και οι δύο χώρες αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα σχετικά με την ε, εφαρμογή της ε, πολιτικής συνοχής και οι υπηρεσίες μας πάντοτε ε, έχουν ως στόχο να αντιπροσωπεύουν και τις, το, το, το, το, μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούμε εκεί. Ξεκινήσαμε το 2013-2014, έχουμε το μεγάλο νοσοκομείο στη Ρήγα, το οποίο ε, ξεκίνησε και στην, ε, στην, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, συνεχίζεται και τώρα και θα επισκεφθείτε και μια σειρά από ενδιαφερόμενους φορείς τον ε, Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Λετωνίας που προτείνει ένα μεγάλο έργο για, την, για τον εξελεκτρισμό του σιδηροδρομικού δικτύου που θα είναι και το μεγαλύτερο έργο αυτής της προγραμματικής περίοδου και ε, αναμένεται να υπάρξει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 347 εκατομμυρίων ευρώ και θα επισκεφθείτε και το Δημόσιο Ίδρυμα Δημόσιας Ανάπτυξης, το Altrum, που είναι η δημόσια τράπεζα που υλοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συστημάτων ενεργειακής αποδοτικότητας της χώρας. Θεωρούμε ότι και οι δύο αυτοί φορείς και οι δύο δικαιούχοι ε, είναι αρκετά αποτελεσματικοί από τη δική μας σκοπιά τουλάχιστον της υπηρεσίας μας και η εφαρμογή του προγράμματος ε, κινείται στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις δαπάνες και ε, ε, με, μεγάλα, ε, με μεγάλη, πολύ καλές αποδόσεις στην επιλογή προγραμμάτων. Δεν βρίσκουμε λοιπόν να υπάρχουν ελλείψεις ή προβλήματα στην περίοδο προγραμματισμού 14-20 και είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή θα σημειώσει και εκείνη την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ε, υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα τα οποία εξετάζουμε βεβαίως και προκειμένου να τα χρηματοδοτήσουμε στο μέλλον αλλά προς το παρόν αυτά θέλω, θέλω να σας πω. Δεν θέλω να σας απαλλάξω ακόμη. Πείτε μας ε, δύο λόγια σας παρακαλώ και για τα έργα. Μιας και είστε εδώ δηλαδή ε, έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε. Παρακαλώ πείτε μας, ενημερώστε μας σχετικά με τα έργα. Ναι βεβαίως καμία αντίρρηση. Τότε θα τα εξετάσω ένα προς ένα τα έργα που θα ε, επισκεφτείτε. Πρώτον, νοσοκομείο της Ρήγας, Στράντιντς, η Πολυκλινική, ε, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, που έχει προσδιοριστεί και ε, στο πλαίσιο του προγράμματος ε, εξυγχρονισμού των υγειονομικών υποδομών της χώρας και Τόσο στην περίοδο του 2007 και στην 2014 ε, η Λετωνία πρότεινε επενδύσεις στο νοσοκομείο αυτό καθώς με, με χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία. Υπήρξε ένα πρώτο έργο μεγάλης κλίμακας στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο με συνολική αξία 46 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε την κατασκευή ενός μεγάλου κτηρίου στο πλαίσιο του νοσοκομείου καθώς και νοσοκομειακό εξοπλισμό. Αυτό το, το έργο έχει ολοκληρωθεί και τώρα προβλέπεται δεύτερη επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία. Περιμένουμε ακόμα την υποβολή της πρότασης για το σχετικό έργο. Δεν έχουμε δει ακόμα το, το, το τελικό ποσό που θα ζητήσει η Λετωνία για την κατασκευή και ενός δεύτερου κτηρίου ε, του νοσοκομείου. Μετά θα πάτε στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Λετωνίας που προτείνει ένα μεγάλο έργο ύψους 441 ε, ε, εκατομμύριων ευρώ με συγχρηματοδότηση και από τα διευθυντικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής συγχρηματοδοτείται και από τη Λετωνία εν, μέρη και μέσω δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που προβλέπει τον εξηλεκτρισμό 300 χιλιόμετρων ραγών σιδηροδρομικών ε, από τα ρωσικά και λευκορωσικά ε, σύνορα ε, προς το κέντρο της, της χώρας, το Ρίσνεσε και στη συνέχεια μέχρι και το λιμάνι της Ρή. αυτή η επένδυση θα διευκολύνει την μεταφορά εμπορευμάτων από τις ανατολικές αγορές και συγκεκριμένα από έναν από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Λετωνίας που είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Κάτι που θα επιτρέψει την ευκολότερη μεταφορά εμπορευμάτων κυρίως προς τα λετωνικά ε, λιμάνια και από εκεί στις σκανδιναβικές αγορές και που θα ε, διευκολύνει την, ε, τη μεταφορά εμπορευμάτων από την Κίνα, την ανταγωνιστικότητα δηλαδή της, ε, της χώρας, γιατί η Λετωνία θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητά της θα βελτιωθεί σε περίπτωση που ο χρόνος μεταφοράς εμπορευμάτων από την Κίνα μειωθεί σε 10 έως 12 ημέρες. Βεβαίως η επένδυση αυτή σχετίζεται και ελέγχεται και με βάση ε, το κριτήριο για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς περιλαμβάνει τη μεταφορά από, το, από τις οδικές μεταφορές στους σιδηροδρόμους. Γι' αυτό και ε, ολοκληρώνουν οι λιτονικές αρχές και μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη βοήθεια του Jaspers, που είναι οι τεχνικές μας υπηρεσίε ε, που ακριβώς θεωρούν ότι αυτή η κοστοποδοτικότητα αυτού του έργου είναι πολύ υψηλή, πολύ θετική. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι το έργο αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια θα επισκεφθείτε το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών και θα παρακολουθήσετε μια πρωτοβουλία που ε, εντάσσεται στην εγγύηση για την απασχόληση των νέων μια διευκόλυνση του κοινωνικού ταμείου που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά για νέους ανέργους και το έργο αυτό, η αξία του οποίου ανέρχεται σε 32 εκατομμύρια και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 19 από το Κοινωνικό Ταμείο και 13 από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, έχει στεφτεί με μεγάλη επιτυχία και θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε και έναν δικαιούχο ε, του Κοινωνικού Ταμείου. Αυτά την πρώτη μέρα, τρίτη μετά το Πάσχα δηλαδή, όταν και θα καταφτάσουμε στη Ρήγα. Μετά θα επισκεφθείτε το Ελληνικό Συνέδριο και την Επιτροπή του Λετωνικού Κοινοβουλίου αρμόδια για τα τα ταμεία που αποτελεί και ένα βήμα όπου συζητούνται τα ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση των νέων. Ε, εκεί λαμβάνονται οι κυριότερες αποφάσεις και τακτικά λαμβάνουν και εκθέσεις από τις ε, διαχειριστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Με άλλα λόγια θα έχετε την ευκαιρία να αποκομίσετε και μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των ε, πολιτικών οργάνων της Λετωνίας. Την επόμενη μέρα το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο. Θα ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί και θα επισκεφθούμε την Altrum, την τοπική τράπεζα επενδύσεων, που ασχολείται με όλα τα ε, χρηματοοικονομικά εργαλεία και από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και την τρέχουσα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την ε, υποστήριξη του προγράμματος των μέτρων ενεργειακής ε, εξοικονόμησης, της ενεργειακής απόδοσης Μιλάμε για κονδύλια που υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πάντοτε χρησιμοποιούνται προς αυτό το σκοπό με προγράμματα χρηματοδότησης για νεοφύης εταιρείε, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία για κεφάλαια κινδύνου και τεχνολογικές ε, εξελίξεις. Το συνολικό ποσό είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρωπαϊκά κονδύλια, το οποίο είναι τεράστιο ποσό για τη Λετωνία. Οι λετωνικές αρχές θα μας πούν ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις, εξαιτία των ευρωπαϊκών δηλαδή κονδυλίων, είναι περίπου πάνω από το 50% των δημόσιων επενδύσεων. Και η συνεισφορά των ευρωπαϊκών κονδυλίων στο ΑΕΠ της χώρας ξεπερνά την ποσοστία μονάδα ετησίως. Το δεύτερο μεγάλο έργο που προωθεί η Altrum είναι το ε, πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια κατοικιών με 130 εκατομμύρια, εκ των οποίων 26 χρηματοδοτούνται από εγγυήσεις και δάνεια για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ενώ τα υπόλοιπα επενδύονται μέσω επιδοτήσεων και δωρεών. Το μείγμα, το επενδυτικό μείγμα, το έχει αποφασίσει η Λετωνία με εξάντε αξιολόγηση των ε, ελήψεων στην αγορά στον τομέα αυτό. Να τονίσω ότι Altum έχει θεωρηθεί ένα κλασικό καλό παράδειγμα ενός ε, σημείου που επιτρέπει να περάσουν όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία ε, μαζί προς την χώρα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει επισημανθεί και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μετά την επίσκεψη αυτή στην Αλτουμ, η αντιπροσωπεία μας θα ταξιδέψει στην πόλη Ολάινε, 100 χιλιόμετρα απόσταση από τη Ρήγα. Με πουλμανάκι θα πάμε. Έχει προβλεφθεί επίσκεψη σε ένα αγρόκτημα τεχνολογικά εξοπλισμένο που έχει πάρει και υποστήριξη από ένα πρόγραμμα στήριξης του ανταγωνισμού. Λέγεται Online Farm με φαρμακευτικά προϊόντα κυρίως. Οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές για τη λετωνική αγορά, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων στη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα έχουμε γύρω στα 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική συμβουλή λοιπόν για αυτή την οφή εταιρεία. Μετά η αντιπροσωπεία θα πάει στην πόλη Μπάλσκα, στο δρόμο προς τα σύνορα με τη Λιθουανία και θα επισκεφθούμε μια εταιρεία παραγωγής τροφίμων που είναι ένας από τους εταίρους του κοινού προγράμματος του Λετωνικού Ερευνητικού Ιδρύματος 5,5 εκατομμύρια περίπου είναι εδώ η συνεισφορά, η συνολική συγγνώμη η συνεισφορά, 3,2 είναι τα ευρωπαϊκά. Υπάρχουν δραστηριότητες για να υποστηριχθεί εξειδίκευση σε αυτήν την μικρή εταιρεία, στην Ομπάλσκα, όπου φαντάζομαι ότι θα δείτε έναν μαχητικό και πολύ δραστήριο τοπικό δικαιούχο. Μετά από αυτό η αντιπροσωπεία θα οδηγήσει με το Πούλμαν ως την Λιθουανία σε ένα διαχειριστικό κέντρο που έχει χρηματοδοτηθεί από από το προηγούμενο διάστημα προγραμματισμού 2007-2013 για ένα σύνολο 11 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο αυτό. Τώρα λειτουργεί αυτό το διαχειριστικό κέντρο. Και το έργο έχει ολοκληρωθεί όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, αν και δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το θέμα. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης προβλέπεται το Πούλμαν, φτάνοντας στο Βίλνιους, να διασχίσει ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο με το λεωφορείο λοιπόν, με το Πούλμαν, που έχει χρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής 84,1 εκατομμύρια ευρώ ήταν ε, το συνολικό κόστος και θα δούμε πώς ακριβώς υλοποιήθηκε. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα προβλέπει επίσκεψη για εργοστάσιο ενέργειας μετά και θα δούμε ποιοι θα συμμετάσχουν. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να έχουμε και λίγες επιπλέον πληροφορίες. Ε, dear Chair, ε, so the, the visit will continue with the Inyalina. Θα συνεχίσουμε με την Ινιαλίνα και από την τελευταία φορά που επισκεφτήκατε την χώρα υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Το θέμα της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι ο στόχος, ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουμε ιδιαίτερα. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι αντιδραστήρες τύπου Τσερνομπίλ έχουν φτάσει πραγματικά στο τελευταίο στάδιο της λειτουργίας τους. Έχουμε νέους κανονισμούς που καθορίζουν πολύ σαφείς ε, ρόλους και διαδικασίες και υπάρχει ένας νέος και βελτιωμένος τρόπος ελέγχου και διαχείρισης αυτών των ε, πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και νέος έλεγχος των προγραμμάτων. Την τελευταία φορά που επισκεφθήκαμε το πρόγραμμα Β1, πρόκειται δηλαδή για την αποθήκευση ε, στο χώρο πυρηνικών ε, αποβλήτων, διαπιστώνουμε και εξάλλου θα επισκεφτείτε αυτό το χώρο στην επισκεφτή σας. Είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε φέτος, στις 25 Φεβρουαρίου, ολοκληρώσει αυτήν την φάση και ότι από την μονάδα 2, από τον αντιδραστήρα της μονάδας 2, έχουν σταματήσει οι δραστηριότητες και παρόλο που αυτό δεν εμπεριέχεται στην ε, προσεχή σας επίσκεψη, είχατε στην προηγούμενη επίσκεψη επισκεφτεί το Β2, 3 και 4, Πρόκειται για τις μονάδες διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών των αντιδραστήρων. Έχουμε και ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχέδιο που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτά είχα να προσθέσω εγώ από δική μα πλευρά. Σα ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι γιατί διαπιστώνω ότι όταν επισκεφτήκαμε την τελευταία φορά ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση και ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Um... Ευχαριστώ. Θα, πιο, θα πω ε, λίγα λόγια για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ESF. E Είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί και αποφέρει ε, αποτελέσματα αλλά και τις συνολικότερες πολιτικές μας Μιλάμε για 32 εκατομμύρια ε, ευρώ στα προγράμματα ESF για 34 μήνες. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό τον Αύγουστο του 2018. Τι αφορά. 7 δυνατότητες προσφορές σε νέους ηλικίας 17 29 ε, ετών ε, από μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες, ανέργους, ε, ακόμη και σε νέους που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης, όπου ξέρετε ότι είναι δύσκολο να παρέχονται στους ανθρώπους αυτούς δεξιότητες και κατάρτιση. Οι νέοι αυτοί λοιπόν θα συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ένα-ενάμιση χρόνο και από εκεί θα αποκτήσουν δεξιότητες, για επαγγέλματα, ε, ε, για έναν κατάλογο που επικυροποιείται κάθε χρόνο ε, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να αποφέρουν και απτά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. Οι νέοι λοιπόν θα συμμετέχουν σε ε, προγράμματα μαθητείας διάρκειας 15 εβδομάδων σε επιχειρήσεις ακριβώς για να αποκτούν ε, πραγματικές εμπειρίες. Αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχος του, του project αυτού. Και το σκεπτικό είναι να δοθούν δεξιότητες σε 6.500 νέους άνεργους έχει επιτευχθεί σχεδόν το 60% του στόχου αυτού. Να προσφερθούν δεξιότητες σε περίπου 1.500 νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων. Εκεί το 80% έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος. Και Επίσης, σκοπός είναι να φτάσουμε και σε 500 νέους στα κέντρα κράτησης. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί στο 100% ήδη. Σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι στους πρώτους έξι μήνες συμμετοχή στα προγράμματα αυτά οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν δουλειά. Το project αυτό είναι ενδιαφέρον πρώτον προφανώς γιατί ακριβώς απευθύνεται σε ανθρώπους που χρειάζονται αυτού του είδους τη στήριξη αλλά και επειδή αποτυπώνει πως τα ταμεία μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολιτικές μας προτεραιότητες. Και υπάρχουν δύο πλαίσια πολιτικής στα οποία θέλω να επιστήσω την προσοχή σας εντός των οποίων εντάσσονται αυτά τα ε, προγράμματα. Πρώτον είναι η εγγύηση για τους νέους που ξεκίνησε το 2014 στη Λετωνία και μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται τρία project. Το ένα είναι αυτό που σας ανέφερα που έχει τον ε, τίτλο επαγγελματική κατάρτιση δεύτερης ευκαιρίας. Δεύτερον, είναι, ε, αφορά τα, τα μέτρα της αγοράς εργασίας και, ε, ε, και ένα άλλο project αφορά τις ανάγκες τους Δήμους. Όλα αυτά έχουν ως στόχο να δώσουν στους νέους ανθρώπους ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία, να επιχορηγήσουν και να επιδοτήσουν μέτρα για την αγορά εργασίας, δίνονται και κίνητρα για την σύσταση και την ίδρυση επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων. Όλα αυτά καλύπτονται λοιπόν από την εγγύηση για τους νέους. Δεύτερος βασικός στόχος αυτής της πολιτικής, εντός του οποίου πρέπει κανείς να ε, εξετάσει όλα αυτά τα project, είναι και η μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματική κατάρτισης στην Λετωνία, είναι ένα ζήτημα ε, στο οποίο έχουν σταθεί και οι συστάσεις ε, αναχώρα. Η Λετωνία λοιπόν μεταρρυθμίζει τα αναλυτικά προγράμματα των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και ανανεώνει συνολικά την ε, εκπαίδευση, την προσέγγιση της ως προς την επαγγελματική κατάρτιση. Αυτά τα project λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και ελπίζουμε στο τέλος να καταλήξουν ε, στο να βρουν οι νέοι άνθρωποι αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη ε, τις δεξιότητες αυτές να βρουν ε, μια θέση απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βόν. Uh, um, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω το γεγονός ότι πήραμε παράταση ε, μία μέρα. Είναι πολύ δύσκολο να επισκεφτείς δύο χώρες σε τρεις μέρες. Τέσσερις λοιπόν καλύτερα είναι. Χαίρομαι που πάμε λοιπόν στη Λιθουανία και στη Λετωνία, σε αυτές τις δύο χώρες που στο παρελθόν δεν έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην πηγαίνουμε μόνο στα μεγάλα κράτη-μέλη αλλά και στα μικρότερα. ακόμη και αν δεν έχουν πάρα πολλά προγράμματα. Είναι, είναι, είναι πάντοτε θετικό και χρήσιμο να παρακολουθούμε τα έργα. Δεν θα σχολιάσω ε, την, ε, τα, τα έργα που θα επισκεφθούμε γιατί είναι δύσκολο πια να αλλάξουν αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε η Κομισιόν για τον εξηλεκτρισμό του συνδρομικού δικτύου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα έργο ε, που δεν έχει χρηματοδοτηθεί επαρκώς ακόμη. Οι προηγούμενες φάσεις χρηματοδότησης έχουν ολοκληρωθεί ήδη, γιατί αν όχι τότε, και βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη φάση υλοποίηση του προγράμματος, τότε δεν θα έχει και ιδιαίτερη αξία η επίσκεψή μας εκεί. Τι ακριβώς δηλαδή περιμένουμε να δούμε ε, ως προς το πρόγραμμα ε, αυτό που αφορά τον αξιλεκτρισμό του συνδρομικού δικτύου. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι το έργο αυτό είναι πολύ καινούριο δεν αποτελεί συνέχεια δηλαδή κάποιου προηγούμενου προγράμματος. Βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας ε, όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία του σχεδιασμού του έργου. Θα μας πούνε λοιπόν ότι θα ανακοινώσουν την ε, προκήρυξη ε, υποβολής προσφορών τον Απρίλιο εξ όσων γνωρίζω και Διοικητικά ε, η αίτηση χρηματοδότησης από τα διευθυντικά ταμεία αναμένεται να καταφτάσει στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το καλοκαίρι. Γιατί επελέγει το έργο αυτό. Φαντάζομαι ότι με δεδομένο ότι πρόκειται για το σημαντικότερο έργο ε, στη Λετωνία, που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην ε, Λετωνία, οι συνάδελφοι προσδιορίσαν το συγκεκριμένο έργο ως πολιτικά σημαντικό έργο που πρέπει να ε, εξεταστεί. Επίσης έχει επισύρει και μια πολιτική συζήτηση στην ε, Λετωνία η οποία οδήγησε σε απόφαση της κυβέρνησης στα τέλη του 2017 σχετικά με την επιλογή της τεχνικής λύσης που θα ε, ε, ε, επιλογή όσον αφορά τη διασύνδεση των ρωσικών και λευκορωσικών συνόρων με την Ρήγα. Υπήρχε και μια άλλη εναλλακτική, να μην συνδεθεί η Ρήγα, αλλά το Πόρτο Βένσκλης στα δυτικά σύνορα της χώρας, το λιμάνι του Βένστης, όπου υπήρχε ε, και εκεί υπήρχαν καλά σημάδια βεβαίως αρχικά κοστοποδοτικότητας, τελικά όμω διαπιστώθηκε ότι θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό και μη βιώσιμο για τον λετωνικό προπολογισμό. Από φυσικής άποψης λοιπόν δεν θα δείτε και πάρα πολλά, αλλά ε, παρόλα αυτά τα στοιχεία που θα λάβετε θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ και έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης και Θέλω να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα ε, για την Volkswagen και κλεισμένο των θυρών 17 και 45 ε, ξεκινάει ε, γι' αυτό πρέπει να απαχωρήσουν όσοι δεν έχουν δουλειά ή θα μείνουν εντός της αιθούσης βεβαίως μόνο όσοι έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη συζήτηση του θέματος αυτού. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν εδώ μαζί μας Χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη Λετωνία. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλώ αποχωρήστε από την αίθουσα. Ευχαριστώ.